κανονισμού με πρώτο θέμα την Καμπότζη και θα δώσω το λόγο στους συντάκτες των ψηφισμάτων. Η κυρία Λόχπιλερ πρώτη. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχουμε εδώ και καιρό μια πολύ αμφιλεγόμενη νομοθεσία για τη ρύθμιση των μη κρατικών ε, ε, των μικροκρατικών οργανισμών στην Γκαμπότζη, ε, τη Λάγκο και βλέπουμε ότι έχει γίνει μια σοβαρή προσπάθεια για την καταπίεση των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Έχουμε να κάνουμε εδώ με την Λάγκο λοιπόν ε, και άλλε απόπειρε εκφοβισμού και παρενόχληση των υπερασπιστών των ανθρωπινών δικαιωμάτων και των εθνικών ε, οργανισμών που δεν μπορούν να λειτουργήσουν, απειλούνται με ποινικά αδικήματα, με ποινικέ κατηγορίες οι οποίες όμως είναι πολιτικά υποκινούμενες. Για άλλη μια φορά βλέπουμε να υπάρχει η Νούσοκα, η Νάιβακα, η Λίμονη και άλλες οργανώσεις, η Τσακρία, ε, που αποκλείονται από την ε, National Election Committee. Διαδηλώσεις, ε, καταστέλλονται από την αστυνομία με διαρκείς παραβιάση των και συλλαμβάνονται και φυλακίζονται οι ακτιβιστές. Εμείς καλούμε την κυβέρνηση Καμπότζης να προχωρήσει στην αποφυλάκηση των κρατουμένων αυτών και να ε, επιτρέψει την ελεύθερη έκφραση της γνώμης. Ε, εδώ μιλούμε για τις αποφάσεις του 2017-2018. Η τα χώριση των ε, ψηφοφόρων επί παραδείγματι και το δικαίωμα ψήφου στους μετανάστες έχει πολύ μεγάλη σημασία και ζητούμε να προχωρήσει σχετική ε, νομοθεσία η ε, κυβέρνηση της Καμπότζης πρέπει να επιτραπεί στην αντιπολίτευση η ελεύθερη πολιτική δράση, οι ηγέτες αντιπολίτευσης αλλά και οπαδοί της υφίστανται διαρκείς απειλές ακόμη και βίαιες επιθέσεις, μέσα στο Κοινοβούλιο ακόμα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κοράου, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Επίτροπε. Μιλάμε για την Καμπότζη Πρόκειται για το τρίτο ψήφισμα σε λιγότερο από ένα χρόνο. Τον Ιούλιο πέρυσι είχαμε κάνει ένα τέτοιο ψήφισμα, μιλώντας ε, για την κατάσταση κατά τον απέναντι μάλλον στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Το πώς αυτό η χώρα ξεπουλιέται στις πολυεθνικές. Και τώρα βλέπουμε πως η κυβέρνηση Ουντσέν είναι μια κυβέρνηση που καταστέλει βία όχι μόνο την ελευθερία έκφρασης και συνέβρεσης, αλλά και οποιαδήποτε μορφή υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξεκινώντας από την περιπόθεση ότι εμείς είμαστε ο βασικός εταίρος της Καμπότζης γιατί έχουμε 410 εκατομμύρια ε, ευρώ που πηγαίνουν ε, προς τα εκεί. Πρέπει ίσως να ξαναδούμε, να επανεξετάσουμε την αναπτυξιακή μας βοήθεια διότι δεν γίνεται να τα στέλνουμε μέσω, με δημοκρατικά, από δημοκρατικές οδούς ιδιαίτερα μέσα στο 2017 εφόσον έχουμε μέσα ας τα χρησιμοποιήσουμε γιατί διαφορετικά θα ξαναβρεθούμε εδώ να λέμε τα ίδια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η επόμενη συντάκτη είναι η κυρία Μακοβέη, την οποία όμω δεν βλέπω στο ημικύκλιο και έτσι δίνω το λόγο στον κύριο Παντσέρη, παρακαλώ. Ένα λεπτό. Όχι, λοιπόν, ο κατάλογος, με συγχωρείτε, έγινε κάποιο λάθος, ε, έχει τώρα τον κύριο Βάιτσενχόλσερ. Ναι, πρόεδρε, με συγχωρείτε, εγώ φταίω γι' αυτό το μπέρδεμα. Λοιπόν, ε, οι τελευταίες εξελίξεις ε, στην Καμπότζη μας ανησυχούν ιδιαίτερα, πάντα στον τομέα των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Πρέπει και πάλι όμως να μιλήσουμε για τα θέματα αυτά. Έχει μια τραγική ιστορία πίσω της η Καμπότζη. Έχει το, τη γενοκτονία των ερυθρών χμέρ των Χμερούς, έχει ένα εμφύλιο ε, πόλεμο, έχει μια θετική εξέλιξη οικονομικά, σε οικονομικούς όρους και θετική πολιτική εξέλιξη στο παρελθόν, με καλές προοπτικές στο παρελθόν και θα μπορούσε το κράτος αυτό πράγματι να προχωρήσει σε μια εξέλιξη αν είχε επιλέξει το δρόμο του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, δυστυχώς υπάρχει ο κίνδυνος, είναι ορατός ο κίνδυνος η Καμπότζη να ξαναπέσει στην αυθαιρεσία και τη διαφθορά. Έχει διέλθει μια συνταγματική κρίση, έγινε μια συμφωνία για μια εκλογική επιτροπή με υποστήριξη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όμως φαίνεται ότι ε, όσο πλησίαζαν οι εκλογές ε, δημιουργούσε περισσότερη νευρικότητα στην κυβέρνηση και έτσι άρχισε η καταστολή έναντι της αντιπολίτευσης και βέβαια ε, να άρχισε να διαχέεται αυτό το κλίμα του φόβου. Εμείς καλούμε την κυβέρνηση της Καμπότης να αφήσει να εγκαταλείψει τον δρόμο αυτό, να αποφυλακίσει όλους τους πολιτικούς κρατημένους και θέλουμε να υπενθυμίσουμε στους Καμποτζιανούς ότι τα σημαντικά μέσα τα οποία διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη χώρα ε, είναι ε, βέβαια πάντα με τον όρο των δημοκρατικών εξελίξεων. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα παρακαλώ τον κύριο Σεκόφσκι που είναι ο επόμενος ο συντάκτης. Κυρίες και κύριοι, το ψήφισμα αυτό είναι μια επίγουσα έκκληση στην κυβέρνηση της Καμπότζης να αλλάξει η κατάσταση στην Καμπότζη, διότι όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, η κατάσταση στη χώρα αυτή χειροτερεύει μήνα το μήνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους μεγαλύτερους ε, εταίρους ε, του βασιλείου της Καμπότζης ε, σε ό,τι αφορά την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε τη σημερινή κατάσταση στη χώρα, όπου δεν έχουμε μόνο καταστολή και καταπίεση της αντιπολίτευσης, αλλά όλων των δημοσιογράφων και άλλοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση της Καμπότζης για να αναγνωρίσει τις δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ, των συνδικάτων και πάνω απ' όλα να δώσει στην αντιπολίτευση τη δυνατότητα να μπορεί να επιτελεί το έργο της, Ιδίω ε, στο πλαίσιο των προεδρικών και τοπικών εκλογών θα πρέπει να φροντίσουμε να διεξάγονται δίκαιες εκλογές και δίκαιες προεκλογικέ εκστρατείες. Εκ μέρους τη δική μου πολιτική ομάδα μπορώ να σα πω ότι θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ στην κατάσταση στην Καμπόντζη και θα φροντίσουμε και εμείς να βοηθήσουμε για τη δίεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών στη χώρα. Η κυρία Βερζία, ευχαριστώ. Τρίτο ψήφισμα πράγματα για την Καμπότζη μέσα σε ένα χρόνο. Πολιτική κρίση από τον Ιούνιο του 2013 καταστολή ε, μέχρι και το συνδικαλιστικό κίνημα είναι θύμα Κυρίως όμως ε, το πρόβλημα που βλέπουμε είναι αρπαγή γεών και σχετικά εγκλήματα. Έχουμε και υπόθεση ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. έχουμε 800.000 θύματα και χιλιάδες, πολλά χιλιάδες θύματα, 60.000 τουλάχιστον το πρώτο μήνα του 2016. Σίγουρα την πρωταρχική ευθύνη την έχουν οι πολυεθνικές και οι ευρωπαϊκές εταιρείες στον τομέα της χλωστοϊφαντουργίας και της ζάχαρης. Οι συνθήκες εργασίας ιδίως για γυναίκες και παιδιά είναι πραγματικά πάρα πολύ ανησυχητικές ανησυχητικέ. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στον τομέα αυτό πρέπει να δράσουμε και να ζητήσουμε αποζημίωση για τα θύματα, αλλά να υπάρξει αναδιαπραγμάτευση συμφωνία όλα εκτό από όπλα. Και να μην εισάγουμε προϊόντα τα οποία είναι προϊόν είτε αρπαγή γεών είτε εκμετάλλευση εργασία. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δούμε ποια είναι η ευθύνη των επιχειρήσεων. Κύριε Επίτροπε. Ωραία είναι να έχουμε εκπρόσωπο τη Κομισιόν, αλλά να μα ακούει τουλάχιστον αυτό ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν. Σα ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ε, έχουμε το θέμα τη ευθύνη των εταιριών. Πρέπει να υπάρχει ένα κατάλληλο νομικό μέσο. Καιρό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να επενδύσουν στο θέμα αυτό. Περιμένω την απάντησή σα. Σα παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής, ο συντάκτης είναι ο κύριος Αουστρεβίτσιος. Ένα λεπτό παρακαλώ. Commissioner colleagues. Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι, πριν δύο μήνε συμμετείχα στην Υποεπιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με, στην αποστολή στην Καμπόζη. Ήταν πολύ ε, συναρπαστική και, και έκθεση στην ε, υποβαθμισμένη πολιτική πραγματικότητα της χώρας. Το πολιτικό κόμμα της αντιπολίτευσης που θα ήθελε να θεσπίσει μια κουλτούρα διαλόγου ε, σταμάτησε μέσω ενός ε, εντάλματος ε, σύλληψης και ένα σωρό ακτιβιστές καταδικάστηκαν ε, για θεμητή και ειρηνική άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης. Εγώ καλώ να την, σε αρχές της Καμπότζη να, καταργήσουν, να, να σταματήσουν αυτές τις συλλήψεις και να αγγιθούν άμεσα την ελευθερία έκφρασης καθώς και όλες τις δημοκρατικές ελευθερίες για τον λαό της Καμπότζη. Καθώ ε, καθώς και να τονίσουμε τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων. Ε, ευχαριστώ πολύ. Και έτσι προχωρούμε, γιατί ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των συντακτών και ακούμε τους ομιλητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Πόψιλα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Άκουσα τους ε, συντάκτες που είπαν πόσο σημαντικό είναι αυτό το ψήφισμα. Και θα ήθελα να το προσυπογράψω και εγώ εκ μέρους της δικής μας πολιτικής ομάδας. Η κατάσταση είναι πιο σημαντική. Ε, ε Ιδίω αν ληφθεί υπόψη τον Ιούλιο, η... ότι θα γίνει η δίκη του Σαν Ρένση σε αυτή τη διαδικασία ε, και απουσία του, ερήμην του θα δικαστεί. Η κυβέρνηση της Καμπότζης δεν πρέπει να συνεχίσει αυτές τις ε, πολιτικά υποκινούμενες βίες επιθέσεις κατά των ηγετών της αντιπολίτευσης. Πολύ καλά ακούσαμε ότι υπάρχει καταστολή των δικαιωμάτων της αντιπολίτευσης, ε, των ε, αντιφρονούν των δημοσιογράφων, καταπιέζονται, τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει και των πολιτών δεν μπορεί να μιλήσει κτλ. Δίνουμε πολύ μεγάλη βοήθεια στη χώρα αυτή. Ε, μήπως αν συνεχίσει αυτή την πολιτική τη θα μπορέσει η Κομισιό να διαθέσει τα, τα χρήματα αυτά για την προσφυγική κρίση για παράδειγμα. Ο κύριος Παντζέρη, ευχαριστώ ε, Πρόεδρε, όπω ήδη υπόθηκε, στην Καμπότζη ακτιβιστέ για τα ανθρωπίνα δικαιώματα μεταξύ των οποίων και ένας υπάλληλο του έχουν κατηγορηθεί για διαφθορά και κινδυνεύουν 5 με 10 χρόνια φυλάκισης. Αυτές οι κατηγορίες πολιτικής ε, προέλευση αποτελούν ανησυχητικά στοιχεία όσον αφορά τη δουλειά αυτών που προσπαθούν να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτή τη χώρα και καθιστούν σαφέ ότι η κυβέρνηση θέλει απλά να βουλώσει στόματα πριν τις επόμενες εκλογές. Ε, διπινική δικαιοσύνη που χρησιμοποιεί του κρατικούς θεσμούς ως μέσα για να ποινικοποιήσει και να τιμωρήσει τις θεμητές δραστηριότητε των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνίας ε, των πολιτών. Αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε είναι απλό και το λέω στον Επίτροπο, πρέπει να αλλάξουμε τη σχέση μας με την Καμπότζη και να θέσουμε συγκεκριμένους όρους. Δηλαδή, το ανθρώπινα δικαιώματα ε, και τα προβλήματα αυτά να αντιμετωπιστούν πραγματικά και αποτελεσματικά. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Νάρτ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ας πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Η Καμπότζη έχει μία διεφθαρμένη ολιγαρχία, μία κλεπτοκρατία που κυβερνά από τον καιρό όπου ο πρώην ε, κόκκινος Χμέρ Χουνσέγκ ε, πέρασε και έφτιαξε τη δική του δικτατορία που βασίζεται σε, στα όπλα και στις ένοπλες ε, δυνάμεις τους, στις ένοπλες ομάδες. Είμαστε μπροστά ενώπιον γκάνγκστερ. Είναι γνωστή η Καμπότζη ως ένας, ε, ως ένας παράδεισος σεξουαλικός στην ουσία, στην πραγματικότητα κόλαση σεξουαλική όπου τα κορίτσια πολλούντες ε, όσους έχουν αρκετά δολάρια για να τις αγοράσουν και η κυβέρνηση κερδίζει από αυτό το ίδιο το σύστημα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να βοηθάμε αυτή την κυβέρνηση διατηρώντας αυτή την κατάσταση στην Καμπότζη και πρέπει να δεσμεύσουμε οπωσδήποτε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια ριζική βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Συναδεινός έχει τώρα το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, δεν γνωρίζω τη γλώσσα της καμπότζης αλλά γνωρίζω πόσο υποκριτές θεωρώ ότι είναι κάποιοι που δήθεν ανησυχούν και ενδιαφέρονται για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην καμπότζη. η έκθεση όπως και τόσες εκθέσεις για χώρες κοντινές ή χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά μας καλεί να καταδικάσουμε την έλλειψη δημοκρατίας την καταπίεση τις πολιτικές διώξεις την καταστολή και την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. υποκρισία αν όχι λαϊκισμός. φυλακή αρχηγού και βουλευτών της αντιπολίτευσης δεν έγινε μόνο στην καμπότζη αλλά και στην ελλάδα. πολιτικές διώξεις αντιπολιτευόμενων κομμάτων συμβαίνουν και στην ευρώπη του κράτους δικαίου εναντίον των εθνικιστικών κομμάτων του front national της lega nord του jobbik του npd. δεν θέλετε να ακούγονται διαφορετικές απόψεις. και πριν βιαστεί κάποιος να με αποκαλέσει ρατσιστή ή απάνθρωπο να απαντήσω μάλλον καλύτερα να καταγγείλω συμπεριφορές μελών της επιτροπής που ασχολείται με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίοι σε εκκλήσεις μου να συζητήσουμε περίπτωση παραβίασης αυτών δεν μπήκαν στον κόπο να απαντήσουν έστω και αρνητικά. ακόμα και ο ίδιος ο πρόεδρος της επιτροπής μόνο ένας απάντησε αναφέροντας ότι για τους επόμενους πέντε μήνες δεν διαθέτει χρόνο είκοσι λεπτών. αν αυτό δεν είναι αντιδημοκρατική συμπεριφορά υποκρισία γελιότητα και ρατσισμός τότε προκαλώ τον οποιονδήποτε να μου δώσει ένα σοφότερο προσδιορισμό. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα οι ομιλητές εξαιδίου ονόματος πρώτα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η πολιτική κατάσταση στην Καμπότζη είναι πολύ σοβαρή και θα χρειαστεί δραστική ε, αντιμετώπιση από τη διεθνή κοινότητα ώστε να προστατευτούν οι ακτιβιστές και οι εκπρόσωποι των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Πρέπει να καταδικάσουμε την καταστολή και ιδιαίτερα θέλω να επισημάνω ότι η Καμπότζη είναι από τα κράτη που κατατάσσονται στο χαμηλότερο επίπεδο Ε, των δημοκρατικών ε, δικαιωμάτων. Ο λαός της Καμπότζης ο ίδιος δεν έχει καμιά εμπιστοσύνη στα δικαστήρια, στη δικαιοσύνη. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μεγαλύτερος χορηγός στην Καμπότζη μπορεί νομίζω να μιλήσει και τη γλώσσα αυτήν. Εάν οι αρχές της Καμπότζης δεν θέλουν να προχωρήσουν σε επικοδομητικό διάλογο με την αντιπολίτευση. Αν δεν καταλαβαίνουν με το καλό, ίσως θα έπρεπε να καταστήσουμε την ε, βοήθεια που προσφέρουμε στη χώρα να την εξαρτήσουμε μάλλον από τις δημοκρατικές εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω τον κύριο Νταϊβιτ Μάρτιν παρόντα στο ε, κοινοβούλιο και στο ημικύκλιο και άρα παρακαλώ την κυρία Χαράνσοβα να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ. Ο Πρωθυπουργό για 30 χρόνια είναι στην εξουσία. Μπορεί να έχουν πάψει αυτές οι σφαγές ε, στους αγρούς ε, που ήταν στο πρόσφατο παρελθόν, όμως ε, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα. Θετικά βήματα έχουν γίνει, αλλά ο Πρωθυπουργός Χαν Κουνσέν θα πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να καταλάβει ότι είναι ένα σύγχρονο κράτος ε, η Καμπότζη και πρέπει να δεχτεί τις δίκαιες ελεύθερες δημοκρατικές εκλογές. Να, υπάρξει, να επιτρέψει ελευθεροτυπία, ελευθερία λόγου και η κυβέρνηση να εργάζεται για όλους τους πολίτες της. Ακόμη και αυτούς που δεν στηρίζουν την σημερινή κυβέρνηση, καταστολή από την κυβέρνηση, επιθέσεις κατά της αντιπολίτευσης, δεν εξυπηρετούν τους στρατηγικούς στόχους της Καμπότζης ή του λαού της. Όταν ήταν εξόριστο στην Κίνα ο τέο βασιλιάς έλεγε ότι απαρνούμε το θρόνο μου για να δείξω στις μάζες ότι δεν υπάρχει κανένας κανόνας διέρη και βασίλευε. Το ίδιο ισχύει νομίζω και για τον Νίν Πρωθυπουργό αλλά και για όλους τους Προέδρους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ε, δεν είμαι σε θέση να δώσω στη διαδικασία καυστεία το λόγο σε όλους, άρα δεν θα ε, λάβουν το λόγο όσοι έχουν ήδη μιλήσει σε προηγούμενη συζήτηση. Ο, από το Ευρωπαϊκό Λέκο Κόμμα, τώρα ακόμα τον κύριο Κουκάν. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Η Καμπότζη είναι κράτος το οποίο ξεκίνησε πριν από μικρό διάστημα ακόμη την ε, οδό της μεταλλαξής, της μεταλλαγής με προσπάθειες αφής από την κυβέρνηση για βελτίωση των συνθήκων στη χώρα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή η κοινωνία, να γίνονται σεβαστές οι θεμελιώδεις ελευθερίες. Σε μια τέτοια περίπτωση λοιπόν ε, παραβιάσεως ή σε τέτοιες περιπτώσεις παραβιάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διώξεων εις βάρος των, ε, της αντιπολίτευσης και των ακτιβιστών δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι και πρέπει να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα τόσο το Κοινοβούλιο όσο και η κοινωνία των πολιτών ε, και πρέπει να υποστηρίξουμε τους αγωνιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα αυτή. Πρέπει λοιπόν να γίνει αυτή η συζήτηση και ε, να προχωρήσει η χώρα προς δημοκρατικές ε, εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ο κύριος Άρνοτ. Πρόεδρε, το εμπόριο και μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη κάποιες χώρες και να τη στηρίξει αν κάπου υστερούν. Μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, οικονομία, ανάπτυξη, εισαγωγές, προϊόντων που δεν μπορούν οι ίδιες οι χώρες να ε, παραγάγουν. Τι πήγε στραβά λοιπόν στην περίπτωση της Καμπαότζης. Αυτό που πήγε στραβά είναι ότι μετετράπει αυτή η ανάπτυξη, αυτή η βοήθεια σε μια κοινική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της χώρας, όπως βλέπουμε ιδιαίτερος από τις ανησυχητικές ειδήσει για τις ε, αρπαγές γεών που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα και ακολουθούν βεβαίως και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι πολιτικοί κρατούμενη, η απουσία δημοκρατίας, οι μασικές καταστρατηγήσεις των δικαιωμάτων. Σε τέτοιες καταστάσεις είναι απολύτως κρίσιμη σημασία να παρακολουθούμε την κατάσταση ώστε η αναπτυξιακή βοήθεια να μην πηγαίνει στα χέρια της κυβέρνησης της Καμπούτζης. Η Πρόεδρος, ε, κύριε Πολτσακ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ήθιστε να συμφωνώ με όλους τους προλαλήσαντες. Είναι κάτι ασυνήθιστο για μένα. Α μην μακρηγορήσω λοιπόν και να πω απλά ότι καταδικάζω τι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη. Ωστόσο, πιστεύω ότι η καταδίκη και η καταγγελία μα θα πρέπει να έχει και έναν πραγματικό αντίκτυπο στι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ με όσου ε, μίλησαν πριν από εμένα και είπαν ότι θα πρέπει και τα μέσα της διπλωματίας να τα χρησιμοποιήσουμε. Παράδειγμα χάρη την χορήγηση αναπτυξιακής βοήθειας. Πρέπει να αντιδράσουμε απέναντι σε αυτή την κατάσταση όπου μια χώρα εξακολουθεί να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. δεν ε, είναι οικονομικά, ε, δεν, δεν εφαρμόζονται οικουμενικά σε όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, βασικά, τα θεμελιώδη δικαιώματα όμως πρέπει να ισχύουν παντού και στην Καμπότζη. Και αν δεν επηρεάσουμε δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση στη χώρα. Έτσι ολοκληρώνουμε τον κατάλογο των αγοριτών και παρακαλώ τον Επίτροπο να λάβει το λόγο. Ε, πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μόλις τον Νοέμβριο κάναμε μια παρόμοια συζήτηση εδώ όσον αφορά την πολιτική κατάσταση στην Καμπότζη. Τώρα, όπως ακριβώς είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, οι ενέργειες αυτής της κυβέρνησης κατά των ε, οργανώσεων των πολιτών ε, προκαλούν σοβαρή ανησυχία. Πρόκειται για διαρκή σοβαρή και παρενόχληση κατά των ηγετών της αντιπολίτευσης ε, παρά την κοινοβουλευτική του ασυλία. Αυτό οδήγησε και στην σύλληψη τεσσάρων υπαλλήλων και ενός πρώην υπαλλήλου της ΜΚΟ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ad Hoc Αυτές οι ενέργειες είναι πολύ ανησυχητικές ε, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της, των εκλογών που προβλέπονται για το 2017 και το 2018 μας αφήγουν με μια ε, αντίληψη περί νέων ε, περιορισμών στην νέα κοινωνία των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κρατήσει σιωπή στη διάρκεια αυτής της περίοδου. Επίσκεψη της αποστολής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 Επίση, έγινε στην ΠΝΟΠΕΜΧ συνεδρίαση, ε, γίνεται κάθε δύο χρόνια και πρόκειται για τα θέματα της συνεργασίας, τη διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο περιθώριο της, συνέλευσης αυτή, της, ε, συνόδου αυτής κάναμε επαφές με τον Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων, οργανώσεις των Νομικιώ και φυσικά με την αντιπολίτευση. Στη διάρκεια όλων αυτών των συνεδριάσεων δε ε, σαφώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε τις σοβαρές ανησυχίες για τη σύλληψη των ε, ε, εκπροσώπων ε, των ΜΚΟ και της αντιπολίτευσης. Καλέσαμε για άμεση απελευθέρωση των υπαλλήλων των ΜΚΟ και αυτό περιλαμβάνεται και στην κοινή δήλωση και στο ε, ανακοινωθέν μετά ο πρεσβευτής μας συνεχίζει να έρχεται σε επαφή με το ε, εκπροσώπους ε, της Καμπότζης και τους πρέσβεις της χώρας και την περασμένη εβδομάδα η κεφαλής της αποστολής της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πνομπέχ εξέδωσαν επίσημη ανακοίνωση καλώντας τις αρχές να πάψουν ε, την δικαστική παρενόχληση και να ε, έρθουν σε επικοδομητικό διάλογο με την αντιπολίτευση. Τόνισαν δε πως πρόκειται για προϋπόθεση για την νομιμότητα των επερχόμενων εκλογών. Ε, είναι δική μας άποψη ε, ότι η κυβέρνηση της Καμπότζης ε, οφείλει να δημιουργήσει και να στηρίξει να διατηρήσει ένα περιβάλλον εντός το οποίο όλα τα πολιτικά κόμματα θα μπορέσουν να αναπτυχθούν χωρίς φόβο για βία ή παρενόχληση. Ε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο ενθαρρύνουμε πολιτική συζήτηση όπου θα ισχύει αμερόληπτα η, ο νόμος, το κράτος δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, από, έχει στηρίξει με 10 εκατομμύρια τις ε, προεκλογικές ε, προσπάθειες και καθώς και την Επιτροπή ε, την ε, πολυμερή για τις εκλογές ε, και βοήθεια παρέχει για την προετοιμασία των επόμενων εκλογών. Είναι σημαντικό να στηρίξουμε την μεταρρυθμιστική διαδικασία μέσω εκλογών. Είναι η μόνη εγγύηση για πραγματικά δημοκρατικές, για δημοκρατική εκλογική αναμέτρηση. Είναι κατά κάποιο τρόπο Ε, μια τέτοια ε, δυνατότητα και ευκαιρία. Βέβαια παρακολουθούμε την κατάσταση σε τακτική ε, βάση. Και ε, θα δούμε ότι ε, θα, θα, πούμε, θα δούμε μάλλον ότι πρέπει να παρατηρήσουμε και τις επερχόμενες εκλογές και σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να, στηρίξει, να στηρίζει μάλλον τις μεταρρυθμίσεις στην Καμπότζη και να ενθαρρύνει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, Επίτροπε. Ε, λάβαμε 7 προτάσεις